αίτηση αναπομπής σε επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 168 της έκθεσης Κόρμπετ σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του κανονισμού. Η εν λόγω αίτηση θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο το βράδυ πριν από την έναρξη της συζήτησης για την έκθεση Κόρμπετ. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η έκθεση της κυρίας Παναγιωτοπούλου Κασιώτου σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.